μερίσες διάταξη. την έκθεση Τσασκόφσκι και Γουαλτιέρη για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη των εκλογών του 2014. Ο πρώτο ομιλητή είναι ο κύριο Τσασκόφσκι. Ένας από τους δύο συνεισηγητέ. Έχετε το λόγο κύριε Τσασκόφσκι. Κυρίε και κύριοι, δεν ήταν εύκολη έκθεση αυτή ιδιαίτερα για όσα κατάγεστε από μεσαίες και μικρότερες χώρες και που ε, πειράζεται ιδιαίτερα από τις προτάσεις που καταθέσαμε στην έκθεσή μας. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να μην ε, αποποιηθούμε των ευθυνών μας. Αποφασίσαμε με τον Ρομπέρτο Γουαλτιέρη να επιλέξουμε μια ρεαλιστική λύση. Ποιε ήταν οι άλλε επιλογέ, να ζητήσουμε περισσότερε έδρε. Αυτό θα ήταν το χειρότερο δυνατό μήνυμα ε, στην σοβούσα κρίση. Και μπορούμε πραγματικά και αξιόπιστα να ζητήσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερε έδρε. Δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν το σωστό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλη λύση ήταν να ζητήσουμε μια ριζική αλλαγή του συστήματος. Αν θέλαμε όμως μια ήπια μετάβαση από τις μικρότερες προς μεγαλύτερες χώρες, ώστε ε, μια και οι μεγαλύτερες χώρες έχουν και περισσότερες ε, ψηφοφόρους που εκπροσωπούν, θα, θα, θα, οδηγούσαμε σε, θα σε μια ριζοσπαστική λύση όπου μερικές χώρες θα έπαιρναν πολύ περισσότερες έδρες και άλλες θα έχαναν περισσότερα από μία. Αλλά τέτοια ριζοσπαστική λύση δεν θα μπορούσε να διδεχθεί ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε και το Συμβούλιο. Αποφάσισαμε λοιπόν ότι προς το παρόν καμία χώρα θα πρέπει να χάσει πάνω από μία έδρα και καμία χώρα δεν θα έπρεπε να κερδίσει έδρες. Μία τέτοια αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο μετά από την αναθεώρηση και άλλων θεσμικών θεμάτων, γιατί η θεσμική μας δομή ε, δράζεται στην ισορροπία μεταξύ του τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο και του τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω ότι μια ριζοσπαστική και ρηξικέλευτη λύση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με άλλες σημαντικές ε, θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως ε, τον τρόπο ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, που δεν είναι καν θέμα συζήτηση αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας υποσχεθώ πάντως ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στο εγγύς μέλλον. Και ίσως τότε, μπορούμε να καταλήξουμε, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα πιο φιλόδοξο. Το σύστημά όμω, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά τις έδρε, προβλέπει την φθήνουσα αναλογικότητα. Ανέκαθεν βέβαια, αντιμετωπίσαμε ένα, δί, ένα δίλημα. Πόσο φθήνουσε και πόσο, αναλογικό θα, πόσο και πόσο αναλογικό θα πρέπει να είναι το σύστημα. Είχαμε την ιστορική εξέλιξη όπου οι μεγαλύτερες ε, χώρες ε, σταδιακά είχαν έδρες, κάτι που απέβει εις βάρος στο σύστημα και αυτό προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε. Επίσης ε, στηριχθήκαμε στην έκθεση Σεβερίν Λαμασούρ, όχι επειδή δεν είναι η καλύτερη έκθεση, αλλά επειδή είχε εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και γι' αυτό το χρησιμοποιήσαμε ως σημείο αναφοράς. Μα ενδιαφέρει η σχέση μεταξύ τη εκπροσώπηση αφενό και του δημογραφικού παράγοντα φετέρου και γι' αυτό προτείνουμε αυτό που λέμε στην έκθεσή μα. Στο σύστημά μα, οι μεσαίε και μικρέ χώρε χώρες υπερεκπροσωπούνται ε, σε ένα αμυγό αναλογικό σύστημα που λαμβάνει υπόψη αυτό που έχει προβλέπει και το Συμβούλιο. Αλλά ένα τέτοιο σύστημα από θεσμική άποψη, από συνταγματική άποψη δεν έχει νόημα. Αντιλαμβάνομαι βέβαια το νόημα των τροπολογιών σας αλλά οι, εισηγητές, οι δεν μπορούμε να δεχτούμε τις τροπολογίες που αφισβητούν είτε, το λογικό, είτε, το, τη λογική είτε την ουσία της έκθεσης. Άλλωστε θεωρώ ότι μας δεσμεύει και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων για να έχει βάρος η απόφασή μας και απέναντι και στο Συμβούλιο θα πρέπει να τη στηρίξει η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια για μερικούς από εσάς δεν θα είναι εύκολο να υπερψηφίσετε την έκθεση, παρόλα αυτά σας ζητώ να συμφωνήσετε με τη συμβαστική μας λύση. Όχι γιατί είναι η, καλή, η ιδεατή συμβαστική λύση, αλλά γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη εφικτή εναλλακτική λύση τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξή σας και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε προς το παρόν τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ευχαριστώ ο κύριος Γουαλτιέρη τώρα, ο δεύτερος συνεισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τσασκόφσκι, ο συνάδελφος συνεισηγητής, μας ε, περιέγραψε πολύ σωστά το στόχο μας. Ε, προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε ένα πολύ λεπτό καθήκον, ε, να τηρήσουμε τη συνθήκη και να λάβουμε υπόψη την ε, προσχώρηση της Κροατίας και την ανάγκη να περιοριστούμε στους 751 ευρωβουλευτές από την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και αυτό θα το κάνουμε με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο. Έχουμε μια αρχή που στηρίζεται στην αρχή της φθήνωσης αναλογικότητας που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και ταυτόχρονα τη χρησιμοποιούμε αυτή την αρχή με ρεαλιστικό και πραγματιστικό τρόπο. Όπως διαπιστώνετε, η πρόταση στηρίζεται σε δύο ασφαλιστικές δικλείδες ε, εφαρμόζει πιστά τις τρεις αρχές ε, που κατοχυρώσαμε με την έκθεση Λαμασούρ Σεβερίν, δηλαδή η μεγαλύτερη χώρα έχει το μεγαλύτερο αριθμό εδρών και μια χώρα από, ένας βουλευτής από μεγάλη χώρα εκπροσωπεί περισσότερους ψηφοφόρους από ότι ο ευρωβουλευτής μικρής χώρας. Και επίση έχουμε και την τρίτη σημαντική αρχή, το ανώτατο και το κατώτατο κατόφλι. 6 τουλάχιστον έδρε και 96 το πολύ. Αποτέλεσμα της πρώτης αυτής φάσης είναι μια σημαντική ε, κατανομή των εδρών, που όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ρεαλιστική ούτε κατάλληλη. Οπότε ε, περνάμε στο δεύτερο στάδιο, που ε, προβλέπει μια πολιτική αντιστάθμιση με βάση τη διπλή αρχή ότι κανένας δεν κερδίζει μια παραπάνω έδρα και κανένας δεν χάνει ούτε μία έδρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ισορροπημένη ε, και από πολιτική άποψη λύση, όπως φάνηκε και από την μεγάλη ε, πλειοψηφία που συγκέντρωσε η πρόταση αυτή στην ε, Συνταγματική Επιτροπή. Γι' αυτό και ευελπιστούμε ότι αντίστοιχη πλειοψηφία θα έχουμε και στην αυριανή ψηφοφορία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η λύση μας είναι η ιδανική λύση. Αλλά είναι τουλάχιστον η λιγότερο ατελής λύση, το μη χείρον μεταξύ των διαφόρων λύσεων. Η αυριανή ε, ψηφοφορία θα δείξει αν η τελευταία έδρα θα παραχωρηθεί από την ε, Σουηδία ή από την Αυστρία, όπως πρότεινε η Συνταγματική οπω προτεινε Είναι ευαίσθητο και λεπτό το θέμα και για τις δύο χώρες. Πάντως το 2014 οι δύο χώρες ε, θα έχουν τουλάχιστον έναν επιπλέον βουλευτή από το 2009. Πάντως η λογική τη της σε δύο φάσει είναι να ζητήσει μια θυσία από τη Σουηδία, ενώ μια... Ε, λογική που προβλέπει μόνο μία φάση θα υιοθετήσει πολύ πιο σφαλμένη λογική. Πάντως, ό,τι απόφαση και λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, χρειαζόμαστε να διασφαλίσουμε την συνοχή και την ισορροπία του συνόλου της πρότασης. Ελπίζω το Συμβούλιο να δεχτεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς τροπολογίες. Γιατί με τροπολογίες ίσως ε, ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ε, του δικαιώματος αρνησικυρίας και έτσι ίσως μας αναγκάσει να μην συμφωνήσουμε με διαφορετικές λύσει από αυτέ δηλαδή που θα απάδουν από το αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορία. Επίσης, είναι σημαντικό και ένα άλλο στοιχείο του ψηφίσματος. Την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προτείνουμε ένα μηχανισμό κατανομή εδρών για τον οποίο χρειάζεται αναθεώρηση των συνθήκων και που θα αντιμετωπίσει το σύστημα και τη ψηφοφορία στο Συμβούλιο και που θα ξανανοίγει το θέμα της ε, εισαγωγή ε, ενός ε, πανευρωπαϊκού ψηφοδελτίου. Είναι σημαντικά θέματα που θα, θα συζητηθούν αργότερα σε μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική θητεία που θα έχει συντακτικό χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως οι προτάσεις αυτές συμβάλλουν στην λύση προς αυτή την κατεύθυνση γι' αυτό και θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους ευρωβουλευτές να την υποστηρίξουν με ζήλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκαζίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για το έργο που έχουν επιτελέσει, που ήταν και δύσκολο και ε, μακροχρόνια. Θα ήθελα να κάνω καταρχάς ένα γενικότερο σχόλιο, με επιτρέπετε. Έχουμε πάρει ένα συγκεκριμένο δρόμο τώρα. Βρισκόμαστε σε μια οδό ε, που οικοδομούμε όλο και περισσότερο στενή ένωση με στόχο ε, την ομοσπονδιακή δομή, διεύρυνση προς άλλες χώρες και πάντα με δημοκρατικές αρχές. Είναι δύσκολο να συνθέσει κανείς όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει το ίδιο ειδικό βάρος στη λύση λήψη των αποφάσεων. Επομένως, κάθε βουλευτής να ε, εκλέγεται από ίσο αριθμό περίπου εκλογέων. Έτσι όμως χάνονται μικρές χώρες και αποκτούν ιδιαίτερο βάρος οι μεγάλες. Γι' αυτό μιλά για φθήνουσα αναλογικότητα η συνθήκη της Λισαβόνας και η Συνταγματική Επιτροπή το ερμήνευσε αυτό. Δηλαδή, ο πληθυσμός της κάθε χώρας θα πρέπει βεβαίως να υπολογίζεται, αλλά να είναι κάπως σταθμισμένη η κατανομή των εδρών με τρόπο δίκαιο. Μας προτείνεται λοιπόν σήμερα μία λύση ρεαλιστική με ελάχιστες θυσίες και ελάχιστα μειονεκτήματα. Θα πρέπει για να χωρέσει η Κροατία να τις κάνουμε λίγο χώρο οι υπόλοιπες χώρες. και να σκεφτούμε και ε, ε, επόμενες ενδεχομένως διευρύνσει. Δεν βρήκαμε λύση εκεί. Είναι σαφές ότι θα πρέπει ο καθένας να συνεισφέρει, να χάσουν κάποιες χώρε έδρες και ταυτόχρονα να σκεφτούμε τι θα γίνει, πώς θα βρεθεί μια λύση ε, τη στιγμή που θα αναθεωρηθούν οι συνθήκες. Δεν θέλουμε τελεσμένα ούτε προσκόμματα στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, η αναθεώρηση των συνθήκων κάποια στιγμή θα κληθεί να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα και γενικότερα ε, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Νομίζω θα πρέπει συλλήφθη να απορριφθούν οι τροπολογίες, έστω και αν ορισμένε είναι ενδιαφέρουσε, και να συμφωνήσουμε με το κείμενο της Συνταγματικής Επιτροπής. Ο κύριος Λάινε. Εξ ονόματο τη Σοσιαλιστική Ομάδα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τι προτάσει του. Είμαστε ένα χρόνο πριν από τι ευρωπαϊκέ εκλογέ και αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που είχαμε να καταλήξουμε σε μια ευρεία πλειοψηφία αύριο στην Ολομέλεια. Η σύνθεση του Κοινοβουλίου πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Η γενική δομή του Κοινοβουλίου ξεκινάει από την εποχή που το Κοινοβούλιο ήταν απλώ ένα συμβουλευτικό σώμα και υπήρχαν τέσσερι κατηγορίες, οι μεγάλε χώρες, οι λιγότερο μεγάλες, οι, πιο μικρές, οι μικρές και οι λιγότερο μικρές. Τώρα που έχουμε το νομοθετικό μα καθήκον, πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και νομιμοποίηση. Χρειαζόμαστε μια νέα φόρμουλα για την καλύτερη εκπροσώπηση των πολιτών τη Ευρώπη στο Κοινοβούλιο μα. Η πρόταση ακολουθεί μια <clears throat> πραγματιστική ε, προσέγγιση. Κανείς δεν χάνει πάνω από ένα βουλευτή και κανείς δεν κερδίζει βουλευτές, είναι λογικό να κάνουμε χώρο για τους νέους συναδέλφους από την Κροατία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε και κάποια λύση για θέματα όπως το αν η Σουηδία ή η Αυστρία θα πρέπει να χάσουν μία έδρα. Αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να υποσχεθούμε είναι ότι μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει και πάλι να επιληφθεί του θέματος αυτού γιατί θέλουμε μία φόρμουλα η οποία θα έχει διάρκεια στον χρόνο και πρέπει να εξασφαλίσουμε και μία καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο πυλώνων της νομοθετικής εξουσίας και πιστεύω και εγώ ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ευρωπαϊκών ψηφοδελτίων, αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε μονάχα μία λύση για το παρόν δεν είναι μία μόνιμη λύση, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή για την πραγματιστική του πρόταση, τους εισηγητές. Ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Στο παρελθόν οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν αντικείμενο παζαριού μεταξύ των κρατών μελών με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα ορθός και δίκαιος. Ιδίω γινόταν αυτό σε, στις τελευταίες στιγμές μιας διακυβερνητικής διάσκεψης. Τώρα όμως χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει το απαραίτητο αυτό έργο το ίδιο και την κατανομή των εδρών. Οι εισηγητές προσπάθησαν να είναι πραγματιστικοί. Βέβαια, ο πραγματισμός δεν αποτελεί την τελειότητα η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων έκανε μια σημαντική τροποποίηση της πρότασής τους υπέρ της Σουηδίας ώστε να μειωθεί ο αριθμός των περιπτώσεων που παραβιάζεται η φθήνουσα αναλογικότητα. Δεν θέλουμε εμείς να ανατρέψουμε στην Ολομέλεια αυτή την <clears throat> αλλαγή και σε πιο μακροχρόνιο επίπεδο η εμπειρία έχει ενισχύσει το επιχείρημα ότι είναι απαραίτητο να βρούμε ένα μαθηματικό τύπο ο οποίος να μπορεί να εφαρμόζεται πριν από κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ένα απλό και διάφανο τρόπο. Πιστεύω ότι αυτή η φόρμουλα θα είναι πολύ κοντά στην λεγόμενη συμβαστική λύση των μαθηματικών του Cambridge που προτάθηκε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πριν από δύο χρόνια. Η έκθεση θέτει αυτό το θέμα και πάλι στην ε, ημερήσια διάταξη της συντακτικής συνέλευσης που ελπίζουμε όταν ξεκινήσει την άνοιξη του 2015 και φυσικά θέτει και το σημαντικό θέμα των υπερεθνικών ψηφοφοριών. Πιστεύω ότι μια συζήτηση για τον αριθμό των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μαζί με μια γενική επανεξέταση των, της στάθμισης των ψήφων <clears throat> στο Συμβουλίο των Υπουργών ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα πραγματικά ισοδίκαιο σύστημα το οποίο είναι απαραίτητο για να υπάρχει μια σωστή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην Ευρώπη. Έχετε πολλά ερωτήματα να αντιμετωπίσετε από δεξιά και αριστερά, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Λάιχτ Φρίντ και μετά η κυρία Φόρντ. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Νταφ, πρέπει να σας πω το εξή. Εγώ δεν σας πιστεύω. Δεν πιστεύω αυτά που είπατε. Μιλάτε για κάποιες αρχές με τα οποία εσείς δικαιολογείτε την απώλεια μιας έδρας για την Αυστρία. Μήπως σκέφτεστε πολιτικά στην περίπτωση αυτή. <coughs> Δεν είναι τυχαίο ότι η Σουηδία έχει πάντα ισχυρή εκπροσώπηση τους φιλελεύθερους, ενώ η Αυστρία όχι. Μήπως αυτό σας αποτελεί το κίνητρό σας. Μήπως είναι λαθασμένο να αντιμετωπίσετε έτσι τα πράγματα. Ελπίζω ότι δεν είναι αυτό το κίνητρό σας, αλλά εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια λογική εξήγηση για το γεγονός ότι η ομάδα σας ζήτησε να αλλάξει την καλύτερη πρόταση των δύο εισηγητών. Μα, λέει ο κύριος Νταφ, εγώ πρέπει με τα να απορρίψω. Α, έχουμε και την κυρία Φόρτ. Η κυρία Βέρτμαν, θέλω να υπενθυμίσω ότι ήρθε ε, πρόσφατα στη φιλελεύθερη ομάδα. <clears throat> θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Φόρτ και μετά θα απαντήσετε και στους δύο ομιλητές ομού, κύριε Νταφ. Φόρτ. Είμαι μαθηματικός και μου αρέσουν οι μαθηματικές απαντήσεις, κύριε Νταφ. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί με τη δική σας πρόταση <clears throat> το Ηνωμένο Βασίλειο έχει λιγότερους βουλευτές κατά κεφαλή από ότι η Γερμανία. Πρώτα απ' όλα λέει ο κύριος Νταφ απορρίπτω κατηγορηματικά και εκφράζω την αποστροφή μου κιόλας για την καταγγελία, την κατηγορία που μου καταλόγησε ο κύριος Λάιτφριντ ότι εγώ είμαι μικροκομματικό στα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πετύχω είναι να έχω μια συνταγματική προσέγγιση, αλλά στο βαθμό που αυτό είναι πραγματιστικά εφικτό. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένας καθαρός μαθηματικός τύπος. Νομίζω και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση. Για να το εξηγήσω. <clears throat> Η διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό μεταξύ της Σουηδίας και της Ουγγαρίας λέει ο κύριος Ντάφ είναι 475.000 άτομα. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή η μικρή διαφορά πληθυσμού αξίζει να μεταφραστεί σε δύο βουλευτές. Η διαφορά μεταξύ της Αυστρίας και της Σουηδίας είναι ένα εκατομμύριο άτομα και εκεί είναι πιο λογικό και δίκαιο να υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των δύο χωρών. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνο για την πληθυσμιακή αύξηση στη Σουηδία ή την Αυστρία ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Απλώς σας ζητώ να δείτε τα αριθμητικά στοιχεία και σε ό,τι αφορά αυτά που είπε η κυρία Φόξ για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ξέρετε, για πραγματιστικούς λόγους δεν προτείνουμε αύξηση στον αριθμό των βουλευτών για οποιοδήποτε κράτος μέλος. Αλλά αν συμφωνήσουμε ένα μαθηματικό πλαίσιο, θα δείτε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία θα έχουν περισσότερους βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Γκέλ Χάφνερ έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ακριβώς αυτή η συζήτηση ότι είχε ταπεινά προσωπικά εθνικιστικά ελαττήρια ένα μέλος της Επιτροπής μας έχει ξαναδίνει και δείχνει πόσο απαραίτητο είναι να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε τακτική. Αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή μας να σταματήσουμε την κατανομή των εδρών μετά από κάθε νέα χώρα που μπαίνει όταν αλλάζει ο πληθυσμός ε, αυθαίρετα να την επαναπροσδιορίζουμε. Χρειαζόμαστε ε, σαφή, ακριβή, διαρκή, βιώσιμη και ε, μονοσήμαντη ε, μαθηματικά φόρμουλα, μαθηματικό τύπο, έτσι ώστε να υπολογίζεται χωρίς καμιά αμφιβολία ο αριθμός των εδρών. Αγωνιστήκαμε γι' αυτό στην Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων, κάναμε μια συμβαστική πρόταση που εγκρίθηκε και επαναλαμβάνω ομόφωνα από το σύνολο της Επιτροπής. Και αν υιοθετηθεί, για αυτή τη φορά ε, θα είναι η τελευταία φορά που προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και στέλνουμε έδρες δεξιά και αριστερά ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τον Ράφαλ και τον Ρομπέρτο ε, που έκανε εξαιρετική δουλειά κατά την άποψή μου, αλλά το θέμα δεν είναι ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στο Συμβούλιο να διαπληκτιζόμαστε για το ποια χώρα θα πάρει πόσες έδρες. Στη δημοκρατία το σημαντικότερο είναι οι κανόνες και ο σημαντικότερος κανόνας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι ε, ο υπολογισμός και η μετατροπή του αριθμού των ε, πολιτών που ψηφίζουν σε βουλευτές για να έχουμε εμεί τη σωστή νομιμότητα και να εκπροσωπούνται όπως τους αναλογεί οι πολίτες. Αυτό θα γίνει τώρα και από την επόμενη φορά θα έχουμε ένα καθαρό μαθηματικό τύπο που θέλουμε σε μια συντακτική συνέλευση να το αποφασίσουμε ε, με φθήνουσα αναλογικότητα, με δικαιοσύνη και προσωπικότητα όλους. Ευχαριστώ. Κύριε Χέφνερ, δέχεστε μια γαλάζια κάρτα. Από το Λόρδο Ντάρτμουθ. Κύριε Χέφνερ, χρησιμοποίησατε τουλάχιστον τρεις φορές τον όρο ομόφωνα στην Επιτροπή σας. Τι θεωρείτε δηλαδή ότι η ομοφωνία μιας Επιτροπής από μόνη της εγγυάται το απάφγασμα της σοφίας όσο και την εγκυρότητα των όσων ψήφισε λόγω επιτροπή. Αγαπητέ συνάδελφοι, ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας, γιατί όντως στην ψηφοφορία ήρθαν κάθε είδους τροπολογίες και μάλιστα εκπροσωπούσαν και εθνικά συμφέροντα ενδεχομένω κάποιες. Και κάποια στιγμή έγινε μια πολύ στενή ψηφοφορία, 11-10 αλλά στο τέλος ήταν ομόφωνη η υιοθέτηση του συνολικού αποτελέσματος. Και θέλω να σας πω ότι εγώ έτσι φαντάζομαι τη δημοκρατία. Και καμιά φορά περιμένω κι εσείς και επιθυμώ να επιδεικνύετε τέτοια στάση και σήμερα στην ψηφοφορία σε ένα κοινοβούλιο μπορεί κανεί να διαπληκτίζεται για διάφορα θέματα, ο καθένα εκπροσωπεί διάφορα συμφέροντα. Αλλά έχουμε ένα κοινό καθήκον. Ακριβώ όταν πρόκειται για εκλογικό δίκαιο και δικαίωμα του κοινοβουλίου να βρούμε κανόνε δίκαιου που να του στηρούν όλοι και εσεί κατά τα άλλα. Και όταν ε, κάποιος παίρνει εδώ το λόγο να μην φωνασκείτε και ενοχλείτε, ε, ε, το Κοινοβούλιο λειτουργεί με δημοκρατικούς κανόνες, έτσι λειτουργεί και η Επιτροπή του και η Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου. Um, την έκθεση αυτή την ετοιμάσαμε προκειμένου να μειώσουμε το μέγεθος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που από 766 θα φτάσουμε σε 766 βουλευτές με την Κροατία από την 1η Ιουλίου. Οι, οι θεώρησαν ότι για να περάσει αυτή η νομοθετική διάταξη στο Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο καμία χώρα πριν της Γερμανίας δεν θα πρέπει να χάσει πάνω από μία έδρα. Και μάλιστα οι συγκητές αποκάλεσαν αυτή τη λύση ρεαλιστική. Και έχουν δίκιο. Δεν είναι βέβαια ιδανική αυτή η λύση. Αλλά αποδέχομαι ότι είναι η πιο πρακτική δεδομένου του στενού χρονοδιαγράμματος που έχουμε για να ε, ανταποκριθούμε στο καθήκον μας εγκαίρως εγκαίρω πριν τι επόμενε ευρωεκλογέ. Εγώ θα προτιμούσα βέβαια ο αριθμό των βουλευτών ε, κάθε χώρα να ανταποκρίνεται στον πληθυσμό τη. Βέβαια, ε, αναγνωρίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση για αργότερα. Δέχομαι τα συμπεράσματα των εισηγητών στην ομάδα μου, παρόλο που δεν θα σας εκπλήσω ότι κάποια από τα μέλη μας δυσαρεστήθηκαν με την έκθεση. Ευχαριστώ κύριος Άγνιου. Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν φαίνεται να χάνει ευρωβουλευτές, η πρόταση αυτή θα πρέπει να καταδικαστεί γιατί υπάρχουν καλύτερα παραδείγματα για το πόσο αντιδημοκρατική, αντιδημοκρατική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα στις διάφορες προτάσεις που εξέτασε η έκθεση κατέληξε να υποβαθμίσει τις μεσαίες και μικρές χώρες. Και μάλιστα ε, γίνεται με πολύ αυταρχικό τρόπο αυτό. Και τελικά δεν έχουν δικαίωμα επιλογής αυτές οι μεσαίες και μικρές χώρες. Και μάλιστα το Συμβούλιο μπορεί να σώσει κάποιες χώρες, αλλά αυτό δεν είναι νομίζω ότι ε, πολύ δημοκρατικός τρόπος. Τώρα ακούμε κάποιες προτάσεις να αναγκάσει το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει τις εκλογές στην Κυριακή και προσπαθεί να του υπαγορεύσει και το πολιτικό περιεχόμενο της εκλογικής, προεκλογικής εκστρατείας. Πώς θα πείσετε ε, τους ε, Βρετανούς ότι είναι ε, δημοκρατικό αυτό το θεσμικό όργανο και όχι μία αντιπροσωπευτική δικτατορία. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Φόξ, τη δέχεστε. Κύριε Άγνιου, μια αντιπροσωπευτικη δικτατορια εχετε μια μπλε καρτα απο τον κυριο φοξ δεχεστε κυριε αγνιου μια στιγμη Ο κύριος Φόξ. Θα ήθελα να πω ότι ε, μετά από αυτό που μας είπε ο κύριος Άγνιου θα ήθελα να μου πει πόσες τοπολογίες κατέθεσε για να βελτιώσει την έκθεση εφόσον την έκρινε τόσο ανεπαρκή. Η παρουσία μου στην ε, Επιτροπή είναι απλώς για να ε, διαπιστώσω τι γίνεται σε εκείνη και να αναφέρω στους Βρετανούς ψηφοφόρους τι γίνεται. Γιατί μερικές φορές το Συντηρητικό Κόμμα συγκαλύπτει τα τεκμενόμενα στην Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Δεύτερη μπλε κάρτα. Κύριε Άγνιο, θα μπορούσατε να συμμετέχετε και στις διαπραγματεύσεις ε, για την έκθεση αυτή. Ήσασταν παρόν σε κάποια από τις ε, διαπραγματευτικές συνεδριάσεις. Ναι, ήμουν σε περισσότερες συνεδριάσεις και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτά που άκουσα. Και μάλιστα σε όλες ε, τις συνεδριάσεις που είμαι παρόν και είμαι στις περισσότερες εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου και τη διαφωνία μου. Ακόμη και όταν είμαι βέβαια, σίγουρα δεν υπερψηφίζω ε, τα επιμέρους σημεία, ούτε και την ε, τελική έκθεση. Είμαι αναπληρωτής βέβαια, δεν έχω απόδειξη ότι, είμαι, θα πρέπει να, ότι ήμουν παρόν, θα πρέπει να τις ε, ψάξω αυτές τις αποδείξεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ υποστηρίζω αυτή την πρόταση για την τροποποίηση σύνθεσης της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι που δεν κάνουν όλε οι πολιτικέ ομάδε. Αλλά σε τρία σημεία θέλω να επικρίνω αυτή την πρόταση. Για μένα δεν είναι σωστό ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει καταφέρει μακροπρόθεσμα να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το πώς γίνεται η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή με το ενιαίο εκλογικό δίκαιο το να πρέπει αυτό να το αποδεχόμαστε σε συνάρτηση με τις ε, έδρες. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα θετικό. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αύξηση ε, δυσφορίας των πολιτών με τις πολιτικές διαδικασίες και κούραση με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πλευρά των πολιτών. Τρίτον, έχουμε ένα γενικό πολιτικό πρόβλημα, όπως είδαμε με την κατανομή των ε, εδρών. Όλοι δρούν έτσι ώστε να μην θυγεί το κράτος μέλος τους. Αλλά οι πολίτες δυσκολεύονται να καταλάβουν ποια διαφορά μεταξύ του Συμβουλίου των Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να έχουμε σαφείς μεθόδους και σαφείς κανόνες ώστε να μπορούμε στο μέλλον να εξασφαλίσουμε και την εσωμάτωση νέων χωρών και να διατηρήσουμε δημοκρατικές συνθήκες. Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια μελλοντική τροποποίηση της σύνθεσης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς μια γενική αναδιάρθρωση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ακόμα και η ισορροπία ε, μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο να επανεξεταστεί και αυτό. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει και οι εκπρόσωποι των πολιτών του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε να θέσετε μια ερώτηση, κύριε Σύμπλα. Σας ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα για τον συνάδελφό μου. Αναφέρθηκε στα πιθανά εθνικά συμφέροντα ότι ο καθένας δεν θέλει να χάσει έδρες. Και εδώ υπήρξε μια καταγγελία κατά του κυρίου Νταφ. Μήπως δείχνει αυτό ότι δεν πρέπει οι ίδιοι οι πολιτικοί να αποφασίζουν πώς εκλέγονται οι πολιτικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μήπως θα πρέπει να γίνεται από άτομα τα οποία είναι έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τα αποφασίζει ένα ανεξάρτητο σώμα, όπως γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος ε, Σόλτς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφασίσουν οι πολιτικοί με δικά τους συμφέροντα. Το θέμα είναι για μένα πόσο σοβαρά παίρνουμε τους πολίτες και τους ψηφοφόρους μας ε, υπόψη μας και στο μέλλον θα πρέπει να εργαστούμε πολύ περισσότερο για να διευκρινίσουμε καλύτερα αυτό το θέμα. Κύριο Σέφλιν. Ο Τζόρτζ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά για το θέμα αυτό. Εκ πρώτης όψεως η ανακατονομή των εδρών δεν θα έπρεπε να είναι πηγή προβλημάτων. Θα έπρεπε να είναι μια αυτόματη συνέπεια της διεύνησης η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνει νέα κράτη-μέλη τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα εκπροσώψης. Η πραγματικότητα, όπως ξέρουμε βέβαια, δεν είναι τόσο απλή. Παρά τις προσπάθειες να γίνει μια τεχνικού χαρακτήρα αναδιανομή με κάποιο μαθηματικό τύπο, η αλήθεια είναι ότι τα πολιτικά δεν μπορούν να εκδιωχθούν από ένα τόσο πολιτικό, πολιτικά φορτισμένο θέμα. Καμιά χώρα δεν θέλει να χάσει έδρες. Οι χώρε αυτέ που χάνουν έδρε λόγω τη διεύρυνση θα κάνουν ό,τι μπορούν για να εξοπλίσουν τι απώλειέ του. Στη συνέχεια υπάρχει το, ρέμα, το θέμα του πώ θα πρέπει να γίνεται καταρχήν η κατανομή των εδρών. Η αρχή τη φθήνουσα αναλογικότητα υπάρχει για να εξασφαλίσει ότι τα μεσαία και μικρά κράτη δεν υποεκπροσωπούνται πολιτικά. Εάν θα γινόταν κάτι τέτοιο, τότε η δύναμή τους, η πολιτική τους φωνή θα ήταν ακόμα πιο αδύνατη από ό,τι είναι τώρα και πρέπει τα μικρά κράτη να τους υπενθυμίσουμε κάθε φορά ότι δεν είναι μονοπόλιο των μεγάλων κρατών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο λοιπόν για να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα δημοκρατικό σώμα να υπάρχει σεβασμός και διαφύλαξη για τα δικαιώματα των μικρών χωρών. Ξέρουμε από την ιστορία της Ευρώπης όταν τα μεγάλα κράτη θεωρούν τα μικρότερα κράτη ως δορυφόρους τους και τα κάνουν ό,τι θέλουν. Οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα της Ευρώπης. Το ίδιο ισχύει και για τις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και η λογική είναι ότι τα περισσότερα κράτη θα πρέπει να χάσουν τουλάχιστον μία έδρα, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να διασφαλιστεί η φθήνουσα αναλογικότητα. Αυτοί που θέλουν να ανατρέψουν αυτές τις δύο βασικές αρχές υποσκάπτουν τη βάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επομένως κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν αντιευρωπαϊκές ε, αντιμετωπίσεις. Κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συνεισφέρω και εγώ στην ευρεία συνένεση και να συγχαρώ τους ηγητές. Εύκολο δεν ήταν, αλλά όπως είπαν και άλλοι έχουν μια λύση ε, βιώσιμη, πραγματιστική για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε εν ώψη και των ευρωεκλογών του χρόνου αλλά επίσης υπόθηκε σωστά ότι είναι προσωρινή αυτή η λύση και το 2015 αναγνωρίζει και έκθεση ότι χρειάζεται κάτι πιο μακροπρόθεσμο, μια λύση που μπορεί να εφαρμόζεται σε κάθε συγκυρία και να μην χρειάζεται διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών ε, και να χάνει μια χώρα, μια έδρα, να την κερδίζει μια άλλη κτλ θα πρέπει να βασίζεται στη φθήνουσα αναλογικότητα όπως ορίζει η συνθήκη. Ένα μαθηματικό λοιπόν σύστημα που να ισχύει κάθε φορά που αλλάζουν τα μέλη του Κοινοβουλίου. Εύκολο δεν θα είναι αυτό το εγχείρημα και ελπίζω η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να αρχίσει νωρί να δουλεύει στην αρχή της επόμενης θητείας. Για να μην ξαναβρεθούμε στα ίδια, να έχουμε δηλαδή μια πραγματιστική λύση μεσοβέζει και ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Παρ' αυτά όσα είπε ο κύριος Άγνου, η σύσταση είναι να γίνουν ευρωεκλογέ 22 ε, με 24 ε, ε, Μαΐου του 2014. Είναι Πέμπτη με Κυριακή αυτό το διάστημα. Δεν απειλείται το Ηνωμένο Βασίλειο που ψηφίζει Πέμπτη. Και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επικυρώσει αυτές τις ημερομηνίε για τις εκλογές. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέχρι να δραστηριοποιηθούν οι δύο εισηγητέ μας. Ε, ήταν σαφή τα πράγματα. Υπάρχει το άρθρο 14.2 για τη φθήνουσα αναλογικότητα ε, και θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ οι τρει αρχέ, γνωστέ σε όλου. Σύμφωνα με του εισηγητέ όμω λέει αυτά δεν είναι μαθηματικά κριτήρια. Ωραία. Α μάθετε μαθηματικά ή να τα ξαναδιαβάσετε. Πραγματικές λύσεις λέτε. Μα αυτά είναι τεχνητές λύσεις, δημιουργήματα που δεν έχουν θεμέλια και είναι εις βάρος μιας χώρας που είναι και πάρα πολύ φιλοευρωπαϊκή. Και θα πρέπει να τιμωρηθεί χάνοντας μία έδρα. δεν μπορούν να αλλάξουν αυθαίρετα ισχύουσε συνθήκες. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά και ελπίζω αύριο να ψηφίσουμε με το σωστό τρόπο και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριο Ζήλε. Ευχαριστώ. Δεν μιλούμε τώρα για μαθηματικά ή για τον αριθμό των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που με απασχολεί είναι οι θεμελιώδεις αρχέ τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Μερικές φορές πίσω από ωραία λόγια όπως συνοχή και αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συγκαλύπτονται ε, εθνικά συμφέροντα μεταξύ ε, συνεισφορέων και δικαιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικές χώρες έχασαν και 10% των, του πληθυσμού τους εξαιτία της κρίσης γιατί μετανάστευσε αυτό σε άλλες χώρες για να βρει δουλειά. Πολλοί, πολλοί συμπολίτε μας εγκαταλείπουν την πατρίδα τους εξαιτία της ανέχειας και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και είδαμε ότι υπάρχουν πολλές διακρίσεις ακόμη και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μερικές χώρες δίνουν ε, μάχη μέχρι τελικής ερανίδος και για την κάθε έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομισματικού Ταμείου ε, και μερικές φορές ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν συζητούμε για το μέλλον μας. Ευχαριστώ κύριο Σμιόλτσερ. Ευχαριστώ πρόεδρε η έλλειπης ε, άμεση αναλογικότητα στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπορεί να οφείλεται στον ειδικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην περιθωριοποιούνται οι μικρές χώρες. Η άμεση αναλογικότητα στην κατανομή των εδρών όμως υπάρχει επιπόλαια κάπως επιφανειακά και ε, αυτό καταλήγει στο να χάνει η χώρα μου ε, μία έδρα, η Αυστρία. Και μάλιστα αυτό φαίνεται αναγκαστικά και λογικό ε, ότι πρέπει να συμβεί. Η Αυστρία δέχτηκε να αυξηθεί κατά ένα τρίτο η δημοσιονομική της επιβάρηση για τους διάφορους μηχανισμούς διάσωσης. Και ο πολίτης στη χώρα μου σιγά σιγά αρχίζει ε, να θεωρεί ότι η παλιά δημοκρατία της Αυστρίας έχει λιγότερο λόγο πλέον αλλά πρέπει να βάζει το χέρι όλο και πιο βαθιά στην τσέπη και οι Αυστριακοί θεωρούν ε, ότι ό,τι αποφασίζεται στην Αυστρία ε, τιμωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές και με κυρώσεις όπως έχουμε ζήσει. Είναι ολέθριο αυτό το μήνυμα και δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι θα αυξηθεί ο ευρωσκεπτικισμός. Γι' αυτό καλώ όλους να δώσουν ένα θετικό μήνυμα στην Αυστρία. Η χώρα πραγματικά καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Ευχαριστώ κύριο Κάρας. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τι δείχνει σήμερα η συζήτηση και μάλιστα σε όλους. Ό,τι χρειαζόμαστε, μια νέα βιώσιμη λύση, ένα μαθηματικό τύπο για την κατανομή των εδρών ε, μετά από προσχώρηση νέων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μιας, διαπαντός χρειαζόμαστε ένα σύστημα διαφανές για τον υπολογισμό της κατανομής των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να μην αρχίσει πάλι αυτός ο καυγάς κάθε φορά που θα έχουμε μια νέα ένταξη. Τι κάνουμε εδώ μία ψήφος σε μία επιτροπή αποφασίζει αν θα έχει μία έδρα περισσότερη ή λιγότερη μία ολόκληρη χώρα. Ωραία, έχουμε ανοίξει τώρα τις ε, θύρες ε, για την εμποροπανήγυρη και το παζάρι. Μπαίνει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται να βρεθούν 11 έδρες. Και υπάρχει και οροφή του αριθμού των εδρών 751. 12 είναι οι χώρες που χάνουν συνολικά έδρες. Αυτή ήταν η πολιτική βούληση, να μην χάσει καμία χώρα περισσότερο από μία έδρα. Ήταν πολιτική βούληση, δεν ήταν μαθηματικός υπολογισμός. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει τις στατιστικές των απογραφών, 8 χώρες θα είχαν χάσει πάνω από μία έδρα και 4 χώρες θα είχαν κερδίσει επιπλέον έδρα. Με αυτό τον υπολογισμό σήμερα η Αυστρία δεν θα έχανε έδρα. Όλοι σήμερα ερχόμαστε και επενούμε τους συζητητές και εγώ ο ίδιος. Ε, τότε γιατί δεν ψηφίζουμε υπέρ της έκθεσης των εισηγητών που τόσο επενούμε. Η έκθεση των εισηγητών ε, εγκρίθηκε ε, και ε, στην Επιτροπή και άλλαξε με μία ψήφο σε μία πρόταση. Εμείς είμαστε υπέρ της έκθεσης προς το παρόν και στο μέλλον να βρεθεί ένας βιώσιμος και διαρκής μαθηματικός τύπος. Ο κύριος Ντάφ, κύριε Κάρες, θέλει να σας θέσει μια ερώτηση. Κύριε Κάρας, σας εκτιμώ ιδιαίτερος, αλλά θα προσπαθήσω να εξηγήσω για ποιο λόγο τροποποίησαμε την έκθεση του εισηγητού. Το κάναμε γιατί παραβίαζε την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Βέβαια, όπως είπα και πριν, δεν μπορούμε να είμαστε πολύ α, σχολαστικοί και να μην αναγνωρίσουμε ότι η συνολική λύση σέβεται αυτή την αρχή. Αλλά φαντάζομαι το δικαστήριο περιμένει ότι θα μειώσουμε τον αριθμό των παραβιάσεων και αυτό τελικά καταφέραμε με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Και ο κύριος Χόκμαρκ, κύριε Κάρας, έχει ερώτηση να σας θέσει. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς, ο κύριος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αγαπητό φίλο Ότμαρ Κάρας ε, κάτι πολύ απλό. Στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων συμφωνήσαμε επί της αρχής ε, επί μιας αρχής που σημαίνει ότι όλες οι χώρες που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανάλογα με το πληθυσμιακό κριτήριο έχουν και συγκεκριμένο ρυθμό βουλευτών. Αυτή την πρόταση ε, συζητούμε τώρα και αυτή θα ψηφίσουμε. Η Αυστρία που είναι η χώρα του κυρίου Κάρας, δεν θέλει να εφαρμοστεί αυτή η αρχή στην Αυστρία, ενώ ισχύει για την Ρουμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και όλες τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αυστρία όμως, που την εκπροσωπείτε εσείς κύριε Κάρες, δεν θέλει αυτός ο κανόνας να ισχύσει για την ίδια. Σας ερωτώ λοιπόν. Γιατί θα πρέπει διαφορά ενός εκατομμυρίου κατοίκων να μην λαμβάνεται υπόψη. Γιατί η Αυστρία έχει ένα εκατομμύριο λιγότερους ε, κατοίκους από τη Σουηδία και διεκδικείται περισσότερου ευρωβουλευτέ από τη Σουηδία. Γιατί θέλετε η Αυστρία να εκπροσωπείται καλύτερα από άλλε χώρε κατά παράβαση του πληθυσμιακού κριτηρίου. Μισό λεπτό η ερώτηση, μισό λεπτό η απάντηση. Δεχτήκατε δύο ερωτήσει, ε, κύριε Κάρα. Έχετε ένα λεπτό για να απαντήσετε. Ναι. Αν με είχατε ακούσει ε, σωστά, κύριε Ντάφ, εγώ δεν επιτέθηκα σε κανένα. Εγώ ζήτησα ε, ένα μόνιμο και διαρκή μαθηματικό τύπο η ερώτηση που μου κάνατε θα πρέπει να απευθυνθεί στους δύο συγητές που σε κάθε βάση υπολογισμού πρότειναν διαφορετική κατανομή εδρών από αυτή που καλούμεθα να ψηφίσουμε τώρα. Και ε, το θέμα δεν, είναι για την Αυστρία, δεν πρόκειται για την Αυστρία. Είναι η βάση υπολογισμού. Δεν είπα τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ότι ήμουν υπέρ της αρχικής έκθεσης. Δεν επιτέθηκα σε κανέναν. Και αυτό που διαμείβεται εδώ μεταξύ μας είναι ακριβώς η έκφραση της κατάστασης ότι χρειαζόμαστε μόνιμους κανόνες. Και η Σουηδία ανέκαθεν ναι, είχε μία έδρα παραπάνω από την Αυστρία, διότι έχουμε διαφορετικό πληθυσμό και με τη νέα κατανομή είχε προταθεί διαφορετικά, όχι όμως επειδή το απαιτήσαμε εμείς, αλλά επειδή έτσι το τεκμηρίωσαν ε, και το αιτιολόγησαν οι, οι Ε, αυτό το ακολουθήσαμε ως πρόταση μας. Ο πρόεδρος. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γιατί αφιέρωσαμε πολύ χρόνο σε αυτό το θέμα. Κυρία Γκυγιόν, παρακαλώ. Oui, Αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θεωρώ ότι η συμβαστική λύση που θα ψηφίσουμε αύριο για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014-2019 δεν μας ικανοποιεί, γιατί η πρόταση αυτή καταλήγει σε ένα αμφισβητήσιμο κείμενο ό,τι αφορά την αρχή της φθήνωσας αναλογικότητας και την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, γιατί έχουμε μια λύση μεν ρεαλιστική, αλλά όχι και ακριβοδίκαιη. Το κείμενο μάλλον, μάλιστα προτείνει για την μελλοντική κατανομή ε, να μην λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα αυστηρά το πληθυσμιακό κριτήριο, κάτι που θα ισχύσει για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Επίσης το κείμενο λέει ότι θα πρέπει στο μέλλον και με αντικειμενικό τρόπο δίκαιο και βιώσιμο και διαφανές ε, να καταλήξει σε μια λύση, κάτι που υπονοεί ότι η τωρινή λύση δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν θεωρώ ότι θα καταλήξουμε συμβεστική λύση για το θέμα αυτό και ούτε θα συγκεντρωθεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Φοβούμαι ε, δυστυχώς ότι δεν ε, θα ευοδοθεί η ρύθμιση αυτή. Ερώτηση του κυρίου Ρανζέλ για την κυρία Γκυγιόμ. Μισό λεπτό παρακαλώ κύριε Ρανζέλ. Κυρία Γκυγιόμ, έχω μία ερώτηση να σας κάνω. Πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε ολόκληρη την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς ε, να αλλάξει τίποτα στο Συμβούλιο. Υπάρχει μια θεσμική ισορροπία. Αυτό που θέλετε είναι να δημιουργήσετε μια ανισορροπία του σχετισμού δυνάμεων και των σχέσεων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αν στο Συμβούλιο δεχτείτε τον ε, Ομοσπονδιακό Κανόνα ε, μία χώρα, μία ψήφος, τότε να δεχτούμε και εδώ τον κανόνα τη αυστηρή αναλογικότητα και να ληφθεί υπόψη και το δημογραφικό κριτήριο. Δεν μπορείτε όμω να έχετε δημογραφικό κριτήριο στο Κοινοβούλιο και όχι στο Συμβούλιο. Αν, ε, αν έχετε χώρε ε, στο Συμβούλιο, θα πρέπει να αναφέρονται οι χώρε και στο Κοινοβούλιο. Ναι, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πρώτον το γεγονός ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της προτινόμενης τώρα λύσης για το εγγύς μέλλον και τις λύσεις για το πιο μακροπρόθεσμο μέλλον. Και είναι κάπως παράδοξο να το τέτοιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Τέιν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ευρωεκλογέ του 2014 είναι πολύ κοντά μας. Θα έχουμε 4,5 εκατομμύρια πολιτών από την Κροατία και έχουμε λόγω της διαφορετικής δημογραφικής ανάπτυξης στα κράτη-μέλη, όλα αυτά μας οδηγούν στην ανάγκη να έχουμε ένα διαφορετικό υπολογισμό για τις ε, έδρες του Κοινοβουλίου. Αλλά είναι ουσιαστικά περιορισμένε οι δυνατότητές μας. Τα μεγάλα κράτη-μέλη υποεκπροσωπούνται και χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν λιγότερου βουλευτέ κατά κεφαλή από ότι η Γερμανία. Οι μικρές χώρες ευνοούνται γιατί έχουν τουλάχιστον ε, πέντε βουλευτές. Τα μικρά, τα μεσαία κράτη-μέλη λοιπόν είναι αυτά τα οποία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουν πάνω από ένα βουλευτή. Γιατί ξέρουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι να χάσουν πάνω από ένα βουλευτή. Και αυτό ε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει δεκτό στο Συμβούλιο, που πρέπει να υπάρξει εκεί μια ομοφωνία για την πρότασή μας. Και μόνο μια τέτοια πραγματιστική λύση μπορεί να δοκιμήσει. Ευχαριστώ κύριο Χεκμάρκ. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση της Συνταγματικής Επιτροπής. Καταρχήν, πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν αριθμό βουλευτών που να εξαρτάται από τον πληθυσμό του. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η αρχή τη σα αναλογικότητα. Όσο πιο πολλού πολίτε έχει ένα κράτο, τόσο λιγότεροι, τόσο περισσότεροι είναι οι πολίτε που εκλέγουν ένα βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώ να εξηγήσω τώρα ότι ένα εκατομμύριο ε, πολιτών περισσότερο δεν υλοποιείται με περισσότερους ευρωβουλευτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κανεί δεν απήντησε σε αυτό το ερώτημα. Η μόνη απάντηση που έχω λάβει στο ερώτημα αυτό είναι ότι το κείμενο ήταν στραβό από την αρχή και επομένω παραμένει στραβό. Και επειδή έτσι πήγε στραβά στην αρχή, πρέπει να εξακολουθήσει να πηγαίνει και τώρα στραβά, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι μα συμφωνούμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, θα πρέπει να το διορθώσουμε και η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων ακολούθησε μια σωστή γραμμή. Αυτό είναι το μόνο που ισχύει. Καταλαβαίνω το πρόβλημα των Αυστριακών ε, Ευρωβουλευτών, αλλά αν δεχθούμε την άποψή της, τότε παραμένει το σύστημα στρεβλό. Γιατί η Αυστρία πρέπει να έχει περισσότερους βουλευτές ε, από τις άλλες χώρες του ίδιου μεγέθους. Γιατί να υπάρξει μια εξαίρεση, μια παρέκκληση για την Αυστρία το μόνο επιχείρημα το οποίο υποστηρίζει την αυστριακή πρόταση και το οποίο στρέφεται κατά τις θέσεις της Συνταγματικής Επιτροπής είναι ότι το σύστημα ήταν στραβό από την αρχή και πρέπει να, να παραμείνει στραβό και τώρα. Μα εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να διατηρούμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Όχι, πρέπει να τα διορθώσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μορέρα, ευχαριστώ. Η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων ε, αποφάσισε να συμφωνήσει με αυτή την ορθολογική λύση για να βρούμε χώρο και για την Κροατία στις επόμενες ευρωεκλογές, ελαχιστοποιώντας ε, τις επιπτώσεις ε, στην γεωγραφική εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προτιμούσα βέβαια να μην χάναμε στη χώρα μου έναν ευρωβουλευτή, αλλά να γνωρίζουμε ότι η λύση είναι ισορροπημένη και βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Στις επόμενες διευρύνσεις θα βρεθούν από άλλες χώρες ε, οι έδρες που απαιτούνται. Επίσης, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση για την ε, μεγάλη γεωγραφική ανακατανομή προτείνεται υπέρ των μεγάλων χωρών ει βάρο τη αρχή τη φθήνου τη αναλογικότητα, που είναι διαφορετική από την αυστηρή αναλογικότητα και θα ήθελα να καταδικάσω αυτή την ε, απόπειρα μερικών συναδέλφων. Οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση τη ίδιας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει και την τροποποίηση του, του τρόπου ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Γιατί δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται η εκπροσώπηση ε, στο Κοινοβούλιο από την εκπροσώπηση στο Συμβούλιο. Όσοι θέλουν να επιφέρουν ρεξικέλευτες μεταρρυθμίσεις στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ανάγκη συσχετισμού στην προσπάθεια αυτή και του Συμβουλίου. Κυρία Βίκστρομ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σωστό και λογικό οι μικρές χώρες με τα ίδια ε, επίπεδα πληθυσμού, με τον ίδιο ρυθμό κατοίκων, να έχουν αντίστοιχες έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε ανέκαθεν διαξυφισμό μεταξύ Αυστρίας και Σουηδίας για το θέμα αυτό. Ξεχνάτε όμως το γεγονός ότι οι Σουηδοί έχουν ένα εκατομμύριο κατοίκους περισσότερους από ό,τι η Αυστρία. Οπότε είναι λογικό και δίκαιο η Σουηδία να κρατήσει τους 20 ευρωβουλευτές της και η Αυστρία να χάσει έναν ευρωβουλευτή, μία έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, ε, κάθε ευρωβουλευτής θα εκπροσωπεί περίπου 475.000 ε, ε, ψηφοφόρους. Αν όμως η Σουηδία χάσει μια έδρα, αν χάσει έναν ευρωβουλευτή, αυτό σημαίνει ότι οι Σουηδοί θα υποστούν διακριτική μεταχείριση θα υποεκπροσωπούνται σε σχέση με τους ε, πολίτες άλλων χωρών. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στην αυριανή ψηφοφορία. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν λάθος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπροκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση μόνο καταρχάς να ευχαριστήσω και τους δύο συγητές ειλικρινά. Ε, δεν έχει φόρο διασκέδασης η δουλειά αυτή. Ε, δεν κερδίζει κανείς, ορισμένοι χάνουν από αυτή τη δουλειά και δεν ε, κερδίζει κανείς μεγάλη συμπάθεια ως εισηγητής για αυτό το θέμα. Και πραγματικά πριτάνευσε μεγάλη λογική και σύνηση και μέθοδος. Ε, και με ένα λογικό τρόπο, εν πάση περιπτώσει, έφεραν σε πέρα σε αυτή τη δουλειά. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, αλλά γενικά είναι μεγάλη συνένεση και ελπίζω να εγκριθεί η πρόταση. Πρέπει να πούμε όμως και το εξής. Είναι μια δίκαιη λύση δεδομένων των συνθηκών, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η μόνη χώρα που δεν χάνει μία έδρα αλλά είναι η Ομοσπονδική Δημοκρατία της Γερμανίας. Και το λέω αυτό μεταξύ σοβαρού και αστείου. Στη συνθήκη της νίκαιας το πουλήσαμε έτσι, αλλά πρέπει να το σημειώσουμε ότι η μοναδική χώρα που χάνει τρεις έδρες είναι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και όλοι οι υπόλοιποι χάνουν μία έδρα. Ας το σημειώσουμε και αυτό. Αν είναι κανείς πρόθυμος εγκαίρος να χάσει τέσσερις έδρες, μετά δεν θα πρέπει να τιμωρείται και γι' αυτό. Ε, ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω, το είπαν και προλαλήσαντες, είναι ότι την άλλη φορά θα πρέπει να κάνουμε γενικότερη συζήτηση που έχει να κάνει με τη δημοκρατική νομιμότητα. Ε, συμφωνώ με εκείνε τις θέσεις που λέγουν ότι η νομιμοποίηση συνδέεται με μια αναλογικότητα. Σε ένα σύστημα ομοσπονδιακό δεν είναι ζήτημα μόνο ενός σώματος. Δεν μπορεί να ορίζεται μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά αυτή η αναλογικότητα, άρα και ε, η εκπροσώπηση θα πρέπει να είναι ένα μείγμα και των δύο σωμάτων. Και εκεί θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση και προς τα έξω και στο συνταγματικό δικαστήριο ότι με τη σημερινή λύση έχουμε πολύ μεγάλη αναλογικότητα σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής ή ε, τη Γερμανία. Θα πρέπει να το ξέρουμε ε, ότι δεν υπάρχει έλλειμμα νομιμοποίησης και δημιουργούμε ε, τις προϋποθέσεις για να δρούμε για τις πολίτες της Ευρώπης και έχουμε και την νομιμότητα και τη δημοκρατία που απαιτείται και την εκπροσώπηση. Ένα λεπτό τώρα η κυρία Μαρίτα Ουλφσκοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγομαι, μάλιστα. Ευχαριστώ έλεγα κύριε Πρόεδρε. Η αρχική πρόταση για την νέα κατανομή των ιδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδυναμώθηκε. Είναι μια ωραία καμπύλη, ε, αλλά αυτή η καμπύλη έχει και μια γωνία, δεν είναι και τα στρογγυλική γωνία, έχει να κάνει με τη Σουηδία. Να σταθούμε λίγο στο παράδειγμα της Σουηδίας. Κανονικά η Σουηδία θα έχανε ένα βουλευτή από τους 20 που έχουμε και αυτό θα σήμαινε ότι σε σύγκριση με την Αυστρία θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Απέναντι σε αυτή την αδικία ε, χρησιμοποίησαμε επιχειρήματα, όχι μόνο εμείς οι Σουηδοί, μας υποστήριξαν και πολλοί άλλοι σε αυτή την προσπάθεια και θέλω να τους ευχαριστήσω η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων άκουσε αυτά τα επιχειρήματα, τα ακολούθησε, πράγμα που με χαροποιεί. Θα παρακαλούσα όλοι να υπερψηφίσουμε τη νέα αυτή πρόταση και να απορρίψουμε την τροπολογία υπαριθμών 8. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα δεν είναι ο καθένας να εκπροσωπεί ίδια συμφέροντα ή να κάνουμε συνταγματική τεχνική και ε, μηχανική. Το θέμα είναι να υπάρχει δικαιοσύνη και δημοκρατία για όλους. Γι' αυτό ελπίζω όλα αυτά τα ωραία που ακούσαμε στη συζήτηση αύριο να ε, βοηθούν στην ψηφοφορία. Τώρα δύο λεπτά η κυρία Κωνσταντς Λεγκρίπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στους δύο συνεισηγητές. Να τονίσω το πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημά τους και τον κατανάγκη ατελή χαρακτήρα της λύσης που έχουν προτείνει αλλά που έχει καταφέρει να πάρει την ευρύτατη υποψήφι, η υποστήριξη της ε, Συνταγματικής Επιτροπής. Είναι μια ρεαλιστική και πραγματιστική λύση, εάν μου επιτρέπετε να πω ότι είναι η μη βέλτιστη λύση. Διατηρεί την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας και προτείνει να μην υπάρξει κανένα κράτος μέλος το οποίο θα χάσει πάνω από μία έδρα. Τούτου λεχθέντος. Πρέπει να πω ότι έχουμε από μια χώρα, την Γαλλία, η οποία μπορεί με θεμητό τρόπο να θεωρήσει ότι υποεκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αντίθετα με άλλα κράτη-μέλη που έχουν υψηλό πληθυσμό, η Γαλλία έχει δημογραφική αύξηση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι πολιτικά εύστοχο και ορθό να να χρησιμοποιεί κανείς την ευκαιρία της ε, έλευσης της Κροατίας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέλευσή μας, ώστε να επιχειρηματολογεί κανείς υπέρ της αύξησης των Γάλλων Ευρωβουλευτών. Κατατέθηκαν τέτοιες τροπολογίες στην Συνταγματική Επιτροπή, τις οποίες εγώ δεν προσυπέγραψα και ευτυχώς απερίθησαν αυτό όμως που είναι σημαντικό για μένα σήμερα και έχω καταθέσει μια τροπολογία προ την κατεύθυνση αυτή που είναι δεκτή στη Συνταγματική Επιτροπή, είναι να πούμε ότι, <clears throat> και θα το πούμε ευθαρσώ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα βγει από τις κάλπες το 2014 θα πρέπει από την αρχή της επόμενης θητείας του να εργαστεί ενδελεχώς το θέμα αυτό για να μπορέσει να καταλήξει σε ένα σύστημα πριν από το τέλος του 2015 που να επιτρέψει μια μόνιμη φόρμουλα αντικειμενικού χαρακτήρα για την κατανομή των εδρών που θα είναι μόνιμη, εξισορροπημένη και αμερόληπτη, που να βασίστε στις δημογραφικές πραγματικότητες. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει σε ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που θα λάβει υπόψη και το λεπτό θέμα της εξισορρόψης των ψήφων στο Συμβούλιο των Υπουργών. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό η κυρία Ρέγνεα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Η έκθεση Τσαρκόφσκι και Γκουαλτιάρη έχουν προτείνει μια εξισορροπημένη λύση ακολουθώντας μια σειρά από αρχές, οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για όλα τα κράτη-μέλη. Να μην υπάρξει διόγκωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να τηρείται η αρχή τη φθήνουσα αναλογικότητα και να υπάρξει μια πραγματιστική αντιμετώπιση. Να μην χάσει κανένα κράτο πάνω από μια έδρα. Η, για την Αυστρία, η απώλεια μια έδρα προ όφελο Σουηδίας σημαίνει ότι μόνο η Αυστρία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση να μην τηρούν οι αρχές και το μπαλάκι για την, ε, τα προβλήματα της Σουηδίας πετάγεται στην Αυστρία. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δεν απαξιαδικία σε βάρος της Αυστρίας και αυτό θα κάνουμε και στην Ορομέλεια, στην ψηφοφορία. Δύο λεπτά για τον κύριο Πάουλου Ρενζέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι η έκθεση αυτή, Ταρκόφσκι και Γκουαλτιέρη, είναι αρκετά εξισορροπημένη και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι πολλές από τις μεσαίες χώρες αποδέχτηκαν το να υπάρξει αυτή η λύση η οποία είναι θετική ακόμα και αν αυτό σημαίνει μια απώλεια εδρών. Εγώ λοιπόν θέλω να συγχαρώ και του εισηγητέ και του εκπροσώπου αυτών των χωρών που δέχτηκαν αυτή την πραγματιστική λύση. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να εξάρω είναι ότι αντίθετα από αυτά που είπε η κυρία Ρέγνερ ή ο κύριος Καράς, η αρχική έκθεση δεν ήταν ορθό. Είχε ένα σφάλμα. Ότι στη σχέση μεταξύ Σουηδία και Αυστρία έβγαινε νικίτρια η Αυστρία. Αυτό σήμαινε ότι παραβίαζε η αυστρια αυτο σημαινει οτι παραβιαζε η αυστρια τα κριτήρια που θεσπίζει η ίδια η έκθεση. Γιατί τονίσαμε όλοι ότι πρέπει να ακολουθούνται αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή των εδρών. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανισότητα ήταν αυτός που προτάθηκε. Και σας λέω και πάλι όλες οι μεσαίες χώρες, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η... το Βέλγιο, η Πορτογαλία κτλ. μπορούν έτσι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει διαφάνεια και ορθολογικός χαρακτήρας στην κατανομή των εδρών. Θέλω να τονίσω και την προσοχή, να φέρω την προσοχή σας σε ένα σημαντικό σημείο, ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ορθή λύση χωρίς να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της στάθμισης των ψήφων στο Συμβούλιο και να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ως ένα σύνολο. Γι' αυτό υποστηρίζω <clears throat> το, αυτά που είπε ο κύριος Μπροκ, αλλά α τα εξηγήσει και στου γερμανού συναδέλφου, του, όπως είναι η κυρία Τούν ότι δεν μπορεί το ΣΑΒ ή η βρεμη να έχουν ε, τρεις ή πέντε ψήφους στην, ε, στο Ευρωκοινοβουλίο εάν τα μικρά κράτη έχουν τόσο μεγάλο ειδικό βάρος στο Συμβούλιο, θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει στα δύο σώματα να υπάρχει μία μορφή ισορροπίας. Λοιπόν, με την έκθεση αυτή αντιμετωπίζουμε το θέμα της Κροατίας, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα της γενικότερης δημοκρατικής εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ένα λεπτό τώρα το λόγο κυρία Ζήτα Ρουγκουρμάη. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Η κατανομή των εδρών είναι ευαίσθητο θέμα. Ήταν ανέκαθεν. Γι' αυτό θα ε, παρότρινα τους συναδέλφους να θετήσουν ε, μια ευρύτερη προοπτική του στόχου της έκθεσης. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να υποδεχθούμε την Κροατία και τους κράτου Ευρωβουλευτές και να προετοιμαστούμε για τις επόμενες ευρωεκλογέ. Η ρεαλιστική προσέγγιση των συνεισηγητών Γουαλτιέρη και Τσασκόφσκι είναι η μοναδική βιώσιμη και εφικτή λύση στο ισχύον πλαίσιο και δεδομένου του στενού χρονοδιαγράμματος. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να τροποποιήσουμε το, το ολόκληρο το σύστημα ανακατανομής χωρίς ε, σημαντικό θεσμικό ανασχηματισμό. Δεν έχουμε ούτε χρόνο, ούτε πολιτική βούληση να πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο πριν τις ευρωεκλογές του 2014. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιτική ισορροπία των θεσμικών οργάνων εξαρτάται όχι μόνο από την ε, κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ε, ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να δούμε και την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στο Συμβούλιο και ούτω καθεξής. Οπότε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν χρόνο να προετοιμαστούν έγκαιρα για τις επόμενες ευρωεκλογέ του 2014, θα ζητούσα από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν την πρόταση των δύο συνεισηγητών. Ευχαριστώ, Ζήτα. Για ένα λεπτό, κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι το βασικό προτέρημα των συνεισηγητών Τσασκόφσκι και Γουαλτέρη δεν ήταν να η ποιότητα της έκθεσης, αλλά το γεγονός ότι έπεισαν την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και ελπίζω ότι αύριο θα πείσουν και την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η λύση τους ήταν η πιο βιώσιμη, πιο ρεαλιστική, πιο συνετή και εφικτή. Η πολιτική τους προσπάθεια ήταν πολύ πιο σημαντική από την μεγάλη ποιότητα και τη μεστότητα της έκθεσής τους είναι επιτακτική ανάγκη να κατανείμουμε τις έδρες και να δώσουμε και στην Κροατία τις έδρες που δικαιούται. Ταυτόχρονα ανοίγουμε και το δρόμο προς το μέλλον, γιατί επισημαίνουμε ότι η ισχύουσα κατανομή δεν είναι ικανοποιητική, ούτε σέβεται πλήρως τις αρχές της αναλογικότητας. Αν και συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκα για την αναλογικότητα και είναι και ασύμετρη κατανομή αυτή ως προς την ε, εκπροσώπηση του Συμβούλιο. Πάντως το πιο σημαντικό είναι ότι με την έκθεση αυτή δεν ε, μεταχειριζόμαστε καμία χώρα, γιατί καμία χώρα δεν χάνει πάνω από μία έδρα. Και από τη στιγμή που υπάρχει συνένεση γι' αυτό, επιβάλλεται η πολιτική λύση και η περισχή της ε, τεχνικής ποιότητας. Γι' αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους συνεισηγητές. Για ένα λεπτό, το λόγο έχει η κυρία Σαντρίν Μπελιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υποτιμώ καθόλου τις προσπάθειες ε, ούτε και το έργο των εισηγητών ε, για την έκθεση αυτή. Αλλά αυτό που προτείνουν για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου το 2014 να μην χάνει ε, κανείς ούτε να κερδίζει περισσότερα από μία έδρα είναι αντίθετο προς την δημοκρατική αρχή που είναι η σωστή εκπροσώπηση και δίκαιη και η ευθύνουσα αναλογικότητα. Τι μας ζητούν σήμερα. Να ψηφίσουμε μια ρεαλιστική πραγματιστική λύση ε, αντιφατική και παρεκκλίνουσα από το πνεύμα της συνθήκης Λισαβόνας. Γιατί ομόφωνα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο καθένα αναβάνει τι ευθύνε του. Δεν είναι δεδομένο αυτό. Εμεί είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κανεί δεν μα υποχρεώνει να κάνουμε εκπτώσει ε, στην εκπροσώπηση από κυβερνήσει που θέλουν ε, το Κοινοβούλιο να μην αντανακλά τη ε, δημοκρατική εξέλιξη στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ε, να συσφίξουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Η συμφωνία αυτή ε, είναι εις βάρος ε, της αξιοπιστίας μας. Θα καταψηφίσω και καλώ τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο. Τελειώσαμε, λέει ο Πρόεδρος και με τους μεμονωμένους βουλευτές. Έχουμε μια σειρά τώρα συναδέλφων που ζητούν το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye. Θα σας διακόπτω ακριβώς επάνω στο λεπτό για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι ή λίγο περισσότεροι από εκείνους που κανονικά δικαιούνται. Ε, πρώτος είναι ο συνάδελφος Σον Κέλλη. Ευχαριστώ. Εμένα μου αρέσουν οι εισηγητές αλλά δεν μου αρέσει η έκθεσή τους. Αυτή η φθήνουσα αναλογικότητα στην πράξη είναι ε, η εκδήλωση δυσαναλογίας. Οι μικρές χώρες, ένα χώρο πριν τις εκλογές δεν ξέρουν πόσους βουλευτές θα έχουν, ούτε πόσες εκλογικές περιφέρειες. Και αυτό είναι η διάκριση κατά των μικρών κρατών ιδιαίτερα. Το 2019 ε, λέτε ε, ε, θα έχουμε βεβαιότητα και μάλιστα τέσσερα χρόνια πριν το 2015. Μα θα πρέπει να κάνουμε προβολές ε, δημογραφικές. Είμαστε η χώρα με την ταχύτερη ανάπτυξη. Τι θα γίνει με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ε, τέσσερις αντί για τρεις βουλευτές θα πρέπει αν είναι αναλογική εκπροσώπηση. Και δεν θα πρέπει να είναι αναχώρα, ανά αριθμό πολιτών που εκπροσωπεί κάθε βουλευτής. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε για να είναι δίκαια. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλήτη. Thank you. I would like to call... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω την ελλαδική κυβέρνηση να θέσει βέτο Ε, από τις 750 έδρες έχουμε μόνο 12. Ε, αυτό είναι υπερέκταση αν θέλουμε να εκπροσωπούμε τα συμφέροντα και να ασχολούμαστε με τις διάφορες υποθέσεις και να παρακολουθούμε στις 22 διαφορετικές επιτροπές τις νομοθετικές διαδικασίες. Θα πρέπει να υπάρχει σταθμισμένη κατανομή για να μπορέσουν να ακούγονται όλοι οι πολίτες. Δεν μπορεί η Γερμανία να έχει 99 έδρες και 12 Ιρλανδία οι μικρές και περιφερειακές χώρες στην Ιρλανδία πώς θα κρατηθούν στην καρδιά της λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη. Καλό την ελλαδική κυβέρνηση να θέσει βέτο για να σταματήσει αυτή η μη δημοκρατική όσο και άδικη κατανομή. Συγγνώμη που σας είπα. Που σας έκανα άντρα, γιατί προφανώς δεν είσαστε. Η κυρία Λούνετσικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως πράσινη και αυστριακή, εγώ κατανοώ για την ανάγκη να υπάρξει μια προσαρμογή λόγω της ένταξης της Κροατίας. Είναι λογικό να υπάρξει λοιπόν μια προσαρμογή, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια γενική λύση η οποία να καλύπτει όλους οι εισηγητές, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα για γενική λύση, κατάφεραν να καταλήξουν σε μια ρεαλιστική ε, συμβαστική λύση, αλλά η οποία περιέχει ακόμα πολλές ανισότητες και ελλείψεις δικαιοσύνης, όπως είπανε και πολλοί συνάδελφοι, καταφέραν να έχουν μια ευρεία πλειοψηφία. Εγώ απέσχα στην ψηφοφορία. Αλλά παραμένουν πολλές ελλείψει δικαιοσύνη και ιδίως, παραδείγματο χάρη, στην περίπτωση μεταξύ της ε, Ουγγαρίας και της, ε, μάλλον, της Αυστρίας και της ε, Σουηδίας. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό έχει νόημα. Την διακόπτει ο πρόεδρος. <clears throat> Δίνω το λόγο στον κύριο Μπάτεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποιητική δικαιοσύνη, το UKIP, να κερδίζει έδρες όλο και περισσότερες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί σε δύο εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθαμε δεύτεροι. Και εμείς θέλουμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πλατφόρμα μας. Σε σχέση με τις εκλογές του 2014 θέλω να κάνω μια πρόβλεψη το, τα το κόμμα το οποίο είναι το πιο πιθανό να έρθει πρώτο στον Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι το UKIP. Αυτό θα καταδείξει και την μεταστροφή πνεύματος των Βρετανών και θα είναι και ένα ορόσημο στο δρόμο να μπορέσει επιτέλους να φύγει η Αγγλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο Ζουάου Φερέρα, κύριο Ζουάου Φερέρα. Α, υπάρχει μία, δεν υπάρχει μπλε κάρτα στο Catch the Eye. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η φέρουσα λογική τη πρόταση κατανομή ε, των αναδρών για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η λογική του φεντεραλισμού. Όχι κυρίαρχων κρατών που είναι ίσα σε δικαιώματα άσχετα με τις διαστάσεις τους, αλλά είναι μια ένωση που την ε, διακυβερνά ένα διοικητήριο που επιβάλλει τη γνώμη τους υπόλοιπους. Επίσης, ε, τιμωρούνται οι μικρές και μεσαίες χώρες προς όφελος των μεγάλων και χώρες όπως η Πορτογαλία χάνουν ε, έδρες και έτσι μειώνεται ακόμη περισσότερο ο πλουραλισμός εκπροσώπησης ε, και απομακρύνεται η Ένωση από την ε, ε, έκφραση πολιτικής, της βούλησης του λαού στις χώρες αυτές. Αυτή είναι μήπως η πρόθεση τελικά, να καταφέρουμε ακόμη ένα πλήγμα στη δημοκρατία. Λάθος είναι αυτός ο δρόμος και με τις, προστά, με τις προτάσεις μας αναζητούμε νέους τρόπους και νέες ε, επιλογές προκειμένου να διαφυλάξουμε τον αριθμό των ευρωβουλευτών των μικρών και μεσαίων χωρών. Η κυρία Σενκλέρ. Ευχαριστώ. Η δημοκρατία είναι ατελής. Βέβαια πιστεύω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τις μικρές χώρες, αλλά η δική μου πατρίδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, υποεκπροσωπείται. Εγώ εκπροσωπώ μια περιοχή, τα West Midlands, με 5 εκατομμύρια κατοίκους. Και στις τελευταίες εκλογές ε, είχαμε 6 ε, ε, δηλαδή εκπροσωπούμε 900.000 και ο καθένας. Ενώ έχουμε ευρωβουλευτές από τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο ε, με 500.000 κατοίκους και επίσης έχουν 6 ευρωβουλευτές. Πώς θα το εξηγήσω αυτό ε, στους ψηφοφόρους μου όταν ένας ευρωβουλευτής από τη Μάλτα και την, το και το Λουξεμβούργο ε, που εκπροσωπεί πολύ λιγότερο κόσμο και από πολύ μικρότερη χώρα ε, έχει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα. Δυστυχώ κλείνει το μικρόφωνο τη κυρία Σενκλέρ. Κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Η λύση που προτείνεται πλήττει κάποιες χώρες όπως τη Ρουμανία. Γίνεται Υπάρχει διάκριση ει βάρο των μικρότερων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προ όφελο των μεγαλύτερων χωρών. Προτιμούμε ένα διαφορετικό σύστημα κατανομής των εδρών μεταξύ των χωρών. Μια τέτοια κατανομή δεν μπορεί να τροποποιείται με μία απλώς προσχώρηση χώρας ε, και τη νέα διεύρυνση να αλλάζουν όλα και να πλήττονται οι παλιές χώρες. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε το σύστημα. Συμφωνούμε με το δημογραφικό κριτήριο. Στην τελευταία απογραφή του 2011 στη Ρουμανία δεν ε, έγινε σωστή και ακριβής ε, απογραφή και φαίνεται ότι ένα εκατομμύριο κάτοικοι δεν περιλήφθηκαν στην απογραφή του 2011. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Κοστέλο. Mr. President. Πρόεδρε, όπως και άλλοι Ιρλανδοί συνάδελφοι, δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτή την έκθεση που προτείνει μείωση των εδρών ε, της Ιρλανδίας για την Κροατία. Είναι κατάφορα αντίθετο με την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Οι μικρές και μεσαίες χώρες υποφέρουν ε, προς όφελος των μεγάλων χωρών. Τι λέει αρχή αυτή, ότι οι χώρες με λιγότερο πληθυσμό θα πρέπει να έχουν ε, πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Η παρούσα πρόταση ε, δεν ε, το εγγυάται αυτό. Η Ιταλία ευνοείται σε σχέση με την Ισπανία. Εμείς χάνουμε μία έδρα και είμαστε ταχύτερα αυξανόμενοι σε πληθυσμό χώρα, ενώ η Φιλανδία και η Σλοβακία έχουν περισσότερο πληθυσμό, χάνουν έδρες. αυτό έχει επιπτώσεις για την αποτελεσματική εκπροσώπηση της Ιρλανδίας, γιατί έχουμε 22 ε, ε, τροπές και είμαστε και περιφερειακή χώρα. Ευχαριστώ κύριος Όπερ Μάιερ. Κύριε Πρόεδρε, με τη χαρμόσυνη έλευση της Κροατίας ε, ξαναμοιράζουμε τις έδρες η Αυστρία χάνει μια έδρα θέλετε υπέρ της ε, Σουηδίας. Με αυτό δεν ευσταθεί ούτε τεκμηριώνεται από την έκθεση. Δεν μπορεί κριτήρια να ορίζονται σε μια έκθεση και μετά αυθαίρετα εις βάρος της Αυστρίας να αλλάζουν. Συχνά ε, οι ε, ε, αφήστανται από τη λογική και είναι λίγο περίεργα αυτά. Πού είναι τα αντικειμενικά κριτήρια ε, θα πρέπει να δούμε τις επιδόσεις τη βαθμολογία των ευρωβουλευτών ε, και οι Αυστριακοί έρχονται πρώτοι. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ γύρω των ομιλητών ε, με τον κύριο Μίτσελ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω πρώτα ότι όλοι μας και εγώ ο ίδιος μιλάμε υπέρ των κρατών μας, ενώ δίνουμε, θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι ε, είμαστε αμερόληπτοι. Δεν μπορεί κανείς να είναι και διάδικος και δικαστής. Λέει η συνθήκη ότι υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός υδρών, εδρών που έχουμε φτάσει και εάν μειώσουμε κατά ένα δωδέκατο τις έδρες των μεγάλων κρατών θα το καταλάβω. Εμείς έχουμε ένα πληθυσμό ο οποίος αυξάνεται αλματοδός και παρόλα αυτά μας αφαιρούν μια έδρα. Δεν νομίζω ότι εδώ πράγματι έχει εφαρμοστεί πράγματι η αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Αυτό μπορεί να τύχει προσφυγής στο Ευρωπαϊκό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κύριε Μίτσελ, έχουμε κλείσει με την οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία και τώρα θα ακούσουμε τους δύο εισηγητές. Ο ένας εκ των δύο έχει καταστεί αόρατο στην αίθουσα, επομένως δίνουμε το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη. Έχετε λοιπόν τέσσερα λεπτά κύριε Γκουαλτιέρη, γιατί μπορείτε να εκπροσωπήσετε και τον συνεισηγητή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν το λόγο στη συζήτηση αυτή και έχουν συμβάλει και πιστεύω επιπλέον ότι έχουν καταδείξει πόσο δύσκολο ήταν το έργο μας ως εισηγητών, συνεισηγητών. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσω του κυρίου Ράγγελ τους βουλευτές από τις χώρες οι οποίες παρά το γεγονός ότι χάνουν μια έδρα μας της πρότασής μας κατάλαβαν τη λογική και τον ορθολογικό χαρακτήρα αυτής της πρότασης και έτσι συνέβαλαν στην θετική απόλυξη της πρώτης φάσης φυσικά μιας διαδικασίας που θα αποδειχθεί σίγουρα δύσκολη και πολύπλοκη. Πιστεύω ότι η συζήτηση κατέδειξε το γιατί είναι δύσκολο το εγχείρημα το οποίο είχαμε να φέρουμε σε πέραση. Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι χρήσιμο να το λέμε όλοι αυτό. Βασίζεται στην αρχή της διτής εκπροσώπησης των κρατών, μελών και των πολιτών η αρχή αυτή γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη από το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό ρεαλιστικά να λειτουργήσουν με δύο βουλές αυτές οι δύο αρχές. Να υπάρχει μία η οποία εκπροσωπεί τα, ένα σώμα νομοθετικό που εκπροσωπεί τα κράτη και ένα που εκπροσωπεί τους πολίτες. Και στα δύο σώματα θα πρέπει να γίνει κάποια διαφορετική μεταρρύθμιση, διαφορετική ρύθμιση των ισορροπιών. Καταλήγουμε λοιπόν σε μια ισορροπία η οποία δεν μπορεί να θεσπιστεί μόνο με ένα αφηρημένο και μονομερή τρόπο, αλλά και είναι και το σωρευτικό αποτέλεσμα μιας ιστορικής διαδικασίας που περιλαμβάνει αντίβαρα και διασταυρούμενες παραχωρήσεις, ώστε να υπάρχει μια στάθμιση στο Συμβούλιο και μια στάθμιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει όλοι να την κατανοήσουν και να κινηθούν σε, στα πλαίσια αυτά με σοφροσύνη. Η κυρία Βέτμαν είπε μια μαθηματική λύση. Μα σας υπενθυμίζω ότι οι μαθηματικές λύσεις που αναφέρονται στην έκθεσή μας θα σημαίνει ότι η Αυστρία θα έχανε τρεις κοινοβουλευτικούς. Η λεγόμενη πρόταση του Κέμπριτς ή η παραβολική λύση ή άλλες μαθηματικές λύσεις. Προσέξτε λοιπόν όταν μιλάτε για τα μαθηματικά, διότι αυτό μπορεί να είναι αρνητικό, να χάσετε. Οι πιο μεγάλες χώρες και οι συνάδελφοι από τις μεγάλες χώρες θέμητα ζητούν να έχουν μια αύξηση στις έδρες τους, αλλά θέλω να τους υπενθυμίσω ότι αυτή η συζήτηση ότι εδώ το πρόβλημα δεν είναι κυρία Μπελιέ η ομοφωνία <clears throat> του Συμβουλίου. Είναι το θέμα της ικανότητας του ίδιου του Κοινοβουλίου να βρει μια λύση και όχι μονάχα να επαφίεται στη δύναμη των πιο μεγάλων που επιβάλλουν τη θέλησή τους στους πιο μικρούς. Χρειάζεται μια όσο δυνατόν ευρύτερη συνένεση. Και νομίζω ότι η αρχή ότι κανείς δεν κερδίζει και κανείς δεν χάνει πάνω από μία έδρα είναι η λιγότερο κακή λύση, η πιο καλή που μπορεί να φανταστεί κανείς. Μπορεί να φαίνεται από μονομερή οπτική γωνία όχι καλή, αλλά αν το δούμε ευρύτερα το γεγονός ότι όλοι εκπροσωπούμε τα κράτη-μέλη μας, θα δείτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μια λύση διαφορετική από αυτήν. Χρησιμοποίησαμε πολλή ώρα σε αυτή τη συζήτηση με το θέμα Σουηδία-Αυστρία. Εγώ έχω κάθε σεβασμό και κατανοώ τις ε, θέσεις που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι και των δύο χωρών. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα λεπτό θέμα, αλλά σας υπενθυμίζω, θέλω να το αποδραματοκοπήσω αυτό το θέμα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και στις ε, δύο περιπτώσεις είχαν και οι δύο, δύο έδρες Ε, παραπάνω καταρχήν και με τον τρόπο αυτό με την πρότασή μας δεν χάνουν πάνω από μία έδρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι συναδέλφοι. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε τα θέματα αυτά από δύο οπτικές γωνίες. Την αρχική πρόταση <clears throat> που είχε σαν στόχο να υπάρξει μία ε, ένα στο ότι η Ουγγαρία χάνει μόνο μία έδρα και όχι δύο ή τρεις <clears throat> και το να υπάρξει κάποια μόνο μία έδρα που παίρνεται από την Σουηδία. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ωραία, ολοκληρώσαμε τη σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την έκθεση της κυρίας Μπόουλς, με θέμα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών. Το λόγο έχει καταρχήν η εισηγήτρια, η κυρία Μπόλς. Παρακαλώ.